Αυτή τη στιγμή περιμένουν 9 άτομα στην Ινδονησία να εκτελεστούν. Δύο Αυστραλοί, ένα Ινδονησίος, δύο Γάλλοι και άτομα άλλης, ε, άλλων εθνικοτήτων. Η, η Ινδονησία μέχρι το φθινόπωρο 2013 είχε ένα μορατόριο στη θανατική ποινή, δεν είχε εκτελέσει καμία θανατική ποινή, έχει αρθεί τώρα αυτό το μορατόμ από το νέο πρόεδρο, ο οποίος απέριψε οποιαδήποτε προσπάθεια να διατηρηθεί το, μοροπα... το μορατόριο αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει τη θανατική ποινή για λόγους αρχής. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και πολλά χρόνια έχουμε ζητήσει να καταργηθεί αυτή η απάνθρωπη μορφή τιμωρίας. Ελπίζω λοιπόν και εξ ονόματος όλων ότι η κυβέρνηση της Ινδονησίας και ο πρόεδρος της Ινδονησίας θα απαρνηθεί την εκτέλεση της θανατικής ποινή και θα επαναφέρει το μορατόριο μου σε σχέση με την εκτέλεση θανατικής ποινής μέχρι ότου καταργηθεί πλήρως και στην Ινδονησία η ποινή αυτή.